ώστε να σταματήσει η εφαρμογή της ανατικής ποινής. Ευχαριστώ την προσοχή σας. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο Κάλλας και τώρα κλείνοντας ε, έχουμε έξι προτάσεις ψηφισμάτων και οι ψηφοφορίες θα γίνουν το τελευταίο θέμα. Επόμενο ζήτημα λοιπόν στην ημερήσια διάταξη, το θέμα της Ουγγάντα, ολοφονία του Ντέιβιντ Κάτο και να δώσω το λόγο στους ε, υπεύθυνου στην Luna ε, Λούνατσεκ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίε και κύριοι. Όλοι μας θα θέλαμε ασφαλώς ο Ντάβιτ Κάτο να μην έχει δολοφονηθεί πριν από κάποιες ημέρες, αλλά όπως και το προηγούμενο Νοέμβριο να βρίσκεται μαζί μας και να συζητάει τις, ε, τα θέματα ε, των ε, δικαιωμάτων και την έλλειψη δικαιωμάτων που έχουν οι ομοφιλόφιλοι και οι λεσβείες στην Ουγγάντα. Όλοι θα θέλαμε να μην είχε πέσει θύμα μια, ενός βίου φόνου, προκειμένου ο Κάτω να μπορούσε να συνεχίσει τη δράση του ως προασπιστής των δικαιωμάτων των λεσβιών, ομοφιλόφιλων, διεμφυλικών και αμφιλοφιλόφιλων στην Ουγγάντα. Χαίρομαι που έχουμε αυτό το ψήφισμα για να καταδικάσουμε την πολιτική ηγεσία η οποία θα επανεκλεχθεί αύριο στην Ουγκάντα. Να καλέσουμε λοιπόν όλες τις δυνάμεις στην Ουγκάντα για να βάλουν ένα τέλος στην, στο μίσος κατά των ατόμων αυτών. Και προκειμένου όλα αυτά τα άτομα, οι λεσβείες, ομοφιλόφιλοι, να μπορέσουν να ζουν ελεύθερα επιτέλους και στην Ουγκάντα. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ευθύνη να προασπίσουμε την ισότητα δικαιωμάτων και στη μνήμη του David Κάτο να συνεχίσουμε τον αγώνα αυτό και στη μνήμη όλων των άλλων ανθρώπων που έχουν χαθεί ε, υποστηρίζοντας τα δικαιώματα αυτών. Γι' αυτό λοιπόν καλούμε την Κάθριν Άστον να προασπίσει ε, τα δικαιώματα αυτά και να χρησιμοποιήσει και το toolkit για τα δικαιώματα των ατόμων αυτών. Ευχαριστώ, συνάδελφε Λούνατσακ. Και τώρα το λόγο έχει για 1,5 λεπτό η Α, και Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε ένα ψήφισμα για το δικαίωμα του ατόμου διαφορετική σεξουαλική προτίμηση στην Ουγκάντα και αλλού. Έγιναν προσπάθειε να εμποδιστεί αυτό που συνέβη στον David Κέιτο. Αυτό ήταν, δραστηριοποιούταν για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δολοφονήθηκε. Θα πρέπει να υπάρχει διάκριση κατά αυτόν τον ανθρώπο σε όλο τον κόσμο, ούτε στην Ευρώπη, ακόμα και εδώ, σε αυτό το σώμα. Ο, ο φόνος του Ντέβιτ Κέιτο είναι δολοφονία, πρέπει να διερευνηθεί διεξοδικά. Οι ένοχοι θα πρέπει να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη και το θέμα των απειλών κατά των ανθρώπων αυτών θα πρέπει να αναλυθεί και να αλλάξει η νοοτροπία. Το Rolling Stone, ένα τοπικό δημοσίευμα και βουλευτέ βουλευτές της Ουγκάντα έπαιξαν ένα ρόλο παρακίνηση αντί να προστατεύσουν του πολίτε. Από όταν δολοφονήθηκε ο David Κέιτο, οι αρχέ σιώπησαν. Η Συμμαχία των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών τη Ευρώπη έθεσε τα δικαιώματα των ανθρώπων αυτών επιτάπητο επανειλημμένα. Και με την υποστήριξη του Κοινοβουλίου παροτείναμε το σεβασμό των ανθρωπίνων του δικαιωμάτων. Διότι ε, για αυτό το πράγμα μιλάμε και δεν θα σιωπήσουμε. Ελπίζω ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καμιά φορά διστάζουν ή δεν θέλουν να υποστηρίξουν τους ομοφιλόφιλους και λοιπά, θα πρέπει να καταλάβουν ότι ποτέ δεν δικαιολογείται ο φόνος ανθρώπου και θα πρέπει να καταδικάζονται αυτά τα φαινόμενα όπως και οι βιοπραγίες κατά άλλων μειονοτήτων σε άλλα μέρη του κόσμου όπως κατά των χριστιανών. Η εξωτερική πίεση τη Ευρωπαϊκή Ενώση να χρησιμοποιήσει την εργαλειοθήκη που έχει στη τη, ούτω ώστε να προωθεί στα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων και στην Ουγγάντα. Ευχαριστούμε στην Αλφέ Σάκε και τώρα ένα λεπτό κύριε Στάνο. Ο φόνος του Ντέβιτ Κάτο είναι αποτέλεσμα εχθρότητα κατά των διαφόρων των ομοφυλοφίλων στην Ουγγάντα. Και κάποιοι βουλευτέ σκληροπυρηνικοί του παρακίνησαν. Δύο φορέ πέρσι καταδικάσαμε τις φρικαλές προσπάθειες που έκαναν κάποιοι βουλευτές στην Ουγκάντα να εγκρίνουν ε, το, την καταδίκη του εγκλήματος ομοφιλοφιλίας όπως το καλείται. Είναι απαράδεκτο να υπάρχει τέτοια μυσαλλοδοξία. Και αυτοί που περασπίζονται βέβαια τα δικαιώματα ομοφιλοφίλων απειλούνται. Αυτό είναι φυσικό και γι' αυτό δολοφονήθηκε ο Ντέβιτ Κέιτο. Ήξερε ότι διέτρεχε κίνδυνο προασπίζοντα του ομοφυλόφιλου δημοσία. Αυτό και άλλοι ομοφυλόφιλοι ε, απεκαλύφθησαν ονομαστικά σε μια εφημερίδα. Βάλαν την φωτογραφία του κάτω από τον τίτλο που, λέει, που έλεγε Κρεμάστε του. Πολλοί στο Λονδίνο ανησυχούν διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει οικονομική βοήθεια σε μια χώρα που τέτοια φρικτά συναισθήματα γίνονται ανεχτά και όχι μόνο και καμιά φορά υποστηρίζονται επίσημα. Ελπίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την προσωπία στο Παναφρικό Κοινοβούλιο θα εξετάσει προσεκτικά ποια δράση μπορεί να λάβει, ούτω ώστε να εκφράσει τη φρίκη μα, τον αποτροπιασμό μα, το θυμό μα για τη δολοφονία του κ. Κέιτο και να υπογραμμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να δίνει βοήθεια στα αφρικανικά κράτη, αλλά θα πρέπει και εκεί να σημειώνεται πρόοδο σε αυτή την ήπειρο όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστούμε στην αδελφή Τάνοκ. Και τώρα η συνάδελφος Βερζιάν για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Βρισκόμαστε στο τρίτο ψήσμα του Κοινοβουλίου ε, από την αρχή της θητείας μας για την ε, κατά των διακρίσεων ε, των λεσβιών, διαφιλικών, ομοφιλόφιλων και φιλομεταβατικών. Ο κύριος κάτω ήταν ε, ένα σύμβολο για την καταπολέμηση της ομοφοβίας στην χώρα του, ειδικά σε ό,τι αφορά την καταδίκη του νόμου Μπατίκ που προχωράει πάρα πολύ στην ε, ποινικοποίηση της ομοφιλοφιλίας που προβλέπει ακόμα και τη θενατική ποινή. Θα πρέπει να, να του απολύσουμε φόρο τιμής, αλλά θα πρέπει επίσης να φροντίσουμε να προστατευτούν αυτοί που κατανομάστηκαν σε, ένα, σε μια φυλάδα. Η στάση λοιπόν των αρχών είναι απαράδεκτη και υποστηρίζεται από τις ακραίες σκεφτικές οργανώσεις. Θα γίνουν εκλογές στην Ουγγάντα ο απερχόμενος πρόεδρος έχει δηλώσει ότι είναι βέβαιος για την επανεκλογή του και ότι θα φυλακίσει όσους τολμήσουν να αφισβητήσουν τα αποτελέσματα των εκλογών. Αυτές οι εκλογές αποτελούν μια ευκαιρία να επενθυμίσουμε στην ε, Ουγγάντα τις υποχρεώσεις του σε θέματα αυτών των δικαιωμάτων και να πούνε ότι οι διακρίσεις, όποιες και αν είναι, ακόμα και αυτές κατά των φιλομεταβατικών, νεφιλικών κλπ, θα πρέπει να γίνουν ε, σεβαστά τα δικαιώματά και τον κύριο Μπανκιμούν να φροντίσει να αγωνιστεί για την αποποινικοποίηση ε, παρόμοιων νόμων και νοοτροπιών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε στην Ανθομυρσιά, αλλά θα ήθελα να επαναλάβω. Εδώ έχουμε ένα λαμπάκι το οποίο να δει όταν ε, πρέπει να πηγαίνει ο μιλητή λίγο πιο σιγά. Ξέρω ότι κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι του οι διερμηνεί, αλλά δεν θα βελτιωθεί οι διερμηνεί όταν διαβάζουν όλο και πιο γρήγορα οι συνάδελφοι σε διπλή ταχύτητα από την κανονική να περιοριζόμαστε στο χρόνο ομιλία που έχουμε και στο περιεχόμενο που χωράει σε αυτό το χρόνο ομιλία για να μπορούν να μεταφράζουν οι διερμηνείς. Ιδάλλως δεν θα καταλαβαίνει κανείς τίποτα παρά μόνο στη γλώσσα σας. Ευχαριστώ. άλλο Κέλλη έχει ένα λεπτό τώρα στη διάθεσή του. Είναι εκτός μικροφώνου και ο Σκέλη. Το θέμα πόσο συνολικό χρόνο αγόρευσης έχουμε, λέει ο Πρόεδρος, δεν είναι στη δική μου εξουσία. Πόσο συνολικός χρόνος διατίθεται για αγόρευσεις. Ε, Κύριε Κέλλη, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, για εκείνους που ζούμε στον ανεπτυγμένο κόσμο, το χάσμα μεταξύ ημών μήτα και των περιοχών των υποσαχαρίων όσον αφορά νοοτροπία και πρακτική είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό. Στην περίπτωση του David Κέιτο βλέπω ένα τέτοιο παράδειγμα. Ήταν ένας άντρα ο οποίος ήταν πατέρας του κινήματος για τα δικαιώματα ε, των ομοφιλοφίλων, ηγέτης του ΣΜΟ που ήταν κίνημα, καταδικάστηκε από ένα δημοσίευμα το Rolling Stone και έλεγε ότι η δίωξη και η εκτέλεση των ομοφιλοφίλων έγινε το περιοδικό να συνεχιστεί και αυτό έγινε 26 Ιανουαρίου τον δολοφόνησαν. Καταδικαστέα καταδικαστές και ο νόμος κατά των ομοφιλοφίλων που δημοσιεύθηκε το 2009 που αν ψηφιστεί πλήρως θα καταδικάζονται οι ομοφιλόφιλοι ε, για 14 χρόνια. Και ακόμα και αυτοί που δεν κατέδωσαν τον ομοφιλόφιλο θα καταδικάζονται για 3 χρόνια. Υπάρχει ελπίδα. Αύριο γίνονται βουλευτικέ και προεδρικέ εκλογέ στην Ουγγάντα. Και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των ομοφιλοφίλων στην Ουγγάντα. Ευχαριστώ και τώρα 1,5 λεπτό έχει το λόγο κ. Κάσμαν. Πρόεδρε, είναι πάντα θλιβερή στιγμή όταν πρέπει να περάσουμε να ψήφισουμε αυτό τον θάνατο ενό προσπιστού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για μένα είναι ακόμα θλιβερότερο, διότι όπω και άλλοι σε αυτό το σώμα τον συνάντησα όταν ήρθε στο Κοινοβούλιο για να απευθύνει η έκκληση ούτω ώστε το Κοινοβούλιο να κινηθεί υπέρ εκείνων που ζουν στην Ουγγάντα σαν αμοφιλόφιλος να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για τον τρόπο με τον οποίο ήταν ενωμένο αυτό το ψήφισμα και είπε ότι το μίσος κατά των ομοφιλοφίλων και των λεσβιών και ο μη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του είναι κάτι απαράδεκτο, τόσο απαράδεκτο. Τι δικαιοσύνη απόδωσαμε εμεί στον Ντέβιτ Κέιτο. Και οι ένοχοι θα πρέπει να σταλούν στη δικαιοσύνη για το φόνο, τον παράλογο φόνο αυτού του νέου αλλά πραγματική δικαιοσύνη μπορεί να αποδοθεί. Σε όλη την Αφρικανική Ήπειρο, όπου όπως είπε και σωστό και ο Στάνοκ, όσον αφορά πολιτικές ελευθερίες και ανθρώπινα δικαιώματα, δώσαμε στους συναδέλφους πάρα πολύ εύκολη ζωή σε αυτά τα ζωτικά θέματα. Ποιο είναι το καλύτερο που απορρέξει από εδώ. Η απεικιοκρατία που επιβάλαμε μέσω των νόμων μας και καμιά φορά μέσω των θρησκειών μας να οδηγήσει στις από ποινικοποίηση σε 38 χώρε τη ομοφιλοφιλίας. Στη Σομαλία, στη Μαυριτανία, στο Σουδάν και στη Βόρεια Νιγηρία επισύρει τη θανατική ποινή η ομοφιλοφιλία. Αν το καταργήσουμε αυτό θα είναι ένα μνημείο όχι μόνο τον Ντέιβιτ Κέιτο που ήταν γίγοντα ανάμεσα στου πυγμέου που διδάσκουν τη δίωξη και τη μυσαλλοδοξία. Θα είναι ένα μνημείο για αυτό το κοινοβούλιο που θα υπερασπίσει εκείνου που δεν έχουν φωνή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, συνάδελφε Κάισμαν. Και τώρα, εξ ονόματος των ομάδων, καταρχάς η κυρία Κρετού έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Και εγώ πιστεύω πως η συζήτηση σχετικά με την παραβίαση των δικαιωμάτων των ε, μειονοτήτων στην ε, Ουγγάντα θα πρέπει να ξεπεράσει την κριτική και θα πρέπει να δούμε τι μέσα έχουμε για να προστατεύσουμε ανθρώπινα δικαιώματα και να δούμε το μέτρο της ε, ευρωπαϊκής διπλωματίας. Έχουμε ψηφίσει και άλλο ψήφισμα για τα δικαιώματα των φιλοφίλων στην Ουγγάντα και για τις διώξεις τους. Πραγματικά αισθάνομαι αποτροπιασμό για την ε, κατάσταση αλλά και για την ε, δισταγμό της επιφυλάξης της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών της να χρησιμοποιήσουν τα μέσα που έχουν διαθεσή τους για να αναγκάσουν τις αρχές της Ουγγάντας να προχωρήσουν σε μια αντικειμενική έρευνα και να παρεμποδίσουν παρόμοιε πράξει στο μέλλον. Ζητάμε λοιπόν από την Κομισιόν μια μεγαλύτερη ανάμειξη στην υπόθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, συνάδελφε Κρατού. Και τώρα η συνάδελφος Στάιν έχει το λόγο για ένα λεπτό. Αξιότιμοι συνάδελφοι, σήμερα θα συζητήσουμε το τρίτο ψήφισμα για το, την ποινική δίωξη της ομοφιλοφιλίας στην Ουγκάντα και θα ψηφίσουμε το σχετικό ψήφισμα και αυτό απειλεί τα δικαιώματα και των νέων. Αυτά αναφέρθηκαν και στο περιοδικό Rolling Stone και ε, καλείται, προκαλείται μίσος εναντίον των ομοφιλοφίλων. Θέλαμε να αποφύγουμε με ένα από τα προηγούμενα ψηφίσματα να παρουσιάζονται τέτοια φαινόμενα βίας. Ε, καταρχάς καλούμε την Ουγγάντα να γίνει αμερόληπτη έρευνα της δολοφονίας του κάτω. Επίσης καλούμε την Ουγγάντα να διώξουν ποινικά ως άτομα ζητούν να εκτελεστούν οι ομοφιλόφιλοι και να αναθεωρήσει η Ουγγάντα επίσης τον νόμο της περί του ομοφιλόφιλους. Ευχαριστώ στον Αλφετάιν και τώρα το λόγο έχει για ένα λεπτό ω στον Συμφωνώ και εγώ με την αγανάκταση που εξέφρασε στην άλλη για τη δολοφονία του Ντέιβιτ Κέιτο. Και αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε τώρα να δείξουμε την αποφασιστικότητά μα. μια σταθερή βούληση για την καταπολέμηση όχι αυτού του μορφής μόνο δολοφονιών αλλά και τι υπερβολές ε, και τι καταδίκες κατά υπό τη μορφή σεξουαλικότητα στην Αφρική. 38 χώρε ε, θεωρείται ως ε, αδίκημα και εμείς πρέπει λοιπόν να το καταπολύσουμε οικονομικά αλλά και πολιτικά διότι θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι πως κατακλείδη μπορούμε να συμβάλλουμε και από οικονομική σκοπιά να καταπολεμήσουμε παρόμοιες καταστάσεις. Είναι απαραίτητο επίση η δίωξη για λόγους γεννητής προσανατολισμού να θεωρηθεί ως απαραίτητο στοιχείο για να, κάνουμε, να παραχωρούμε το καθεστώς του πρόσφυγα στα άτομα αυτά τα οποία δεν μπορούν να ζήσουν πλέον στις χώρες τους. Εάν δεν το πράξουμε τώρα, στο μέλλον θα θρυνήσουμε και άλλα θύματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ στον Αλφαρμέ και τώρα ο συνάδελφος Τσαρνέσκη για ένα λεπτό. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι η τρίτη φορά που συζητάμε τη χώρα αυτή σε μία περίοδο λίγων μηνών. Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Συμφωνώ με τους ε, προηγούμενους ομιλητές. Δεν μιλάμε μόνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα μίας ομάδας ανθρώπων. Όχι. Το θέμα είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα εν γέννη, αλλά ασφαλώς και οι μειονότητες πλήττονται ιδιαίτερα και είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες και βάλλοντες. Νομίζω ότι η φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να ακουστεί ξανά και ξανά. Αυτό είναι ουσιώδου σημασία και χαίρομαι που όλε οι πολιτικέ ομάδε μιλούν με μία φωνή παρά το γεγονό ασφαλώ ότι τονίζουν ενδεχομένω διαφορετικέ πτυχέ του θέματο ανάλογα με τον προσανατολισμό τη καθεμία. Επίση θα πρέπει να προστατεύονται τα άτομα διαφορετικού γενετήσιου προσανατολισμού. Θα πρέπει να υποστηρίζονται να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής και στην πολιτική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα το λόγο, μάλλον τώρα θα πάρουν το λόγο η συνάδελφος Έστιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο φόνος του David Κέιτο, ενός από τους πιο γνωστούς προσπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουγγάντα, είναι απόρρια του μίσου. Μίσου κατά των ομοφυλόφιλων. Ακόμα και αν ο δολοφόνο τελικά προσαχθεί στη δικαιοσύνη, η ατμόσφαιρα μίσου θα παραμείνει και θα επιβεβαιωθεί και από τους νόμους που προβλέπουν διακρίση. 38 χώρες στην Αφρική ποινικοποιούν, έχουν ποινικοποιήσει την ομοφυλοφιλία σε τέσσερι χώρες, μάλιστα, τιμωρείται με θαντική καταδική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τον εκδημοκρατισμό των αφρικανικών χωρών. Πόσο αίμα πια πρέπει να χυθεί, πόσοι άνθρωποι πρέπει να πεθάνουν προτού η διεθνή κοινότητα αναγκάσει αυτές τις χώρες να αλλάξουν την νομοθεσία τους. Θα πρέπει να εξετάσουμε και τον ρόλο της Εκκλησίας. Αντί να προωθεί την αγάπη προς αλλήλους, προωθεί το μίσος, διακηρύττοντας ότι η ομοφυλοφιλία είναι μια ασθένεια προσίαση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα θα αναφέρετε ότι οι μη εγγυγραμμένοι μπορούν να πάρουν το λόγο για ένα λεπτό παραπάνω. Το λόγο έχει η κυρία Σινκλέρ, λοιπόν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σημειώσω ένα διαδικαστικό. Είναι η τρίτη φορά που μας είχατε υποσχεθεί χρόνο αγόρευση και δεν μα είχατε δώσει χρόνο. Επειδή είμαστε μία κυκραμένη δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε και δικαίωμα να μιλήσουμε. Και τώρα θα ξεκινήσω την ομιλία μου. Θα ήθελα να, να ξεκινήσω, να αποτίσω φορό τιμή στον ε, David Κάτο για το έργο του στην Ουγγάντα. Γιατί δεν προσπίστηκε μόνο τα δικά του δικαιώματα, αλλά και τα δικαιώματα όλων των ατόμων με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό στην Ουγκάντα αλλά και στην υπόλοιπη Αφρική. Είναι λυπηρό ότι ήρθε σε αυτό το κοινοβούλιο τον προηγούμενο Οκτώβριο και παρόλα αυτά δεν ακούσαμε τις προειδοποιήσεις του ούτε τη διεθνή κοινότητα και τώρα έχει χαθεί, δολοφονήθηκε. Είναι απίστευτο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα παρέχει βοήθεια προς την Ουγκάντα και ελπίζω ότι μετά τις εκλογές θα αναθεωρήσουμε την βοήθεια αυτή σε περίπτωση που δεν θα δοθεί αμνηστία σε άτομα που έχουν διαπράξει εγκλήματα ως προς ε, τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους. Ένα τελευταίο στοιχείο. Είναι πολύ λυπηρό που η τρέχουσα Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ουγγρική Προεδρία, αποφάσισε να απαγορεύσει ε, ένα γκέι πριν τον Ιούνιο. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, συνάδελφε Σινκλέρ. Συνάδελφε Σίνκλερ, ναι, ε, συγγνώμη, σας μιλώ, σα μιλώ, λέει ο Μου αναφέρετε από τους υπαλλήλου σας ότι δεν αναφέρθηκε ο χρόνος αγορευσή σα Να σας πω προσωπικά ότι αν οι υπάλληλοι σα έχουν προβλήματα, ναι, τι να κάνουμε, πρέπει να βάλετε και τα ακουστικά σας. Θα σας τα πω κατευθείαν με... Θα το, προσε... προσέξω εγώ προσωπικά. το... Κοιτάξω εγώ προσωπικά. Εν πάση περιπτώσει, ο συνάδελφος Σιλβέστρη στην διαδικασία κάτω διάει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η καταδίκη του Κέιτο χρειάζεται να καταδικαστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι αυτό είναι μόνο ένα επεισόδιο του ευρύτερου προβλήματο των διακρίσεων που υπάρχουν ανά τον κόσμο κατά των μειονοτήτων πολιτιστικών, εθνικών, εθνοτικών, ε, θρησκευτικών. Πριν από μερικέ εβδομάδε ε, ψηφίσαμε ένα κατεπήγον ψήφισμα καταδικάζοντα αυτό το οποίο συνέβησε στου κόπτε χριστιανού στην Αλεξάνδρεια τη Αιγύπτου που δολοφονήθηκαν μόνο και μόνο γιατί ήθελαν να εκφράσουν την πίστη του ε, ανοιχτά. Η Ουγκάντα είναι μια χώρα ιδιαίτερα ευαίσθητη και ευάλωτη. Έχει γίνει αντικείμενο ε, από διάφορες πολυεθνικές εταιρείες. Θα πρέπει λοιπόν η Ουγκάντα σήμερα να τύχει της προσοχής της Ευρώπης μέσω της ικανότητές μας να προάγουμε την δημοκρατία και τα ε, πολιτικά δικαιώματα σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφε Σιλβέστρης και τώρα στην συνάδελφος για και για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το μίσο και η παραβιάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά των σεξουαλικών μειονοτήτων εξακολουθούν να υπάρχουν σε όλο τον κόσμο και τα πρόσφατα νέα για την ολοφονία του κυρίου Ντέβιτ κάτω στην Ουγγάντα αποτελεί ένα ακόμα λυπηρό παράδειγμα της βίας που αντιμετωπίζουν τα άτομα αυτά. Η δολοφονία του κυρίου Κάτω θα πρέπει να διερευνηθεί. Και όλοι οι υπεύθυνοι θα πρέπει να προσαχθούν στη δικαιοσύνη. Αναφέρθηκε ότι κάποιες αρχές, όπως για παράδειγμα η εφημερίδα Rolling Stone, ζήτησαν δημόσια τη δολοφονία του David Κάτω. Θα πρέπει να διερευνηθούν καταλήλως αυτές ε, οι κατηγορίες. Να πω, Πρόεδρε, ότι μου προκάλεσαν φρίκι ε, οι δηλώσεις του Υπουργού Ηθικής και Δοντολογίας ε, της Ουγκάντα, μιλώντας για τους ομοφιλόφιλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, συνάδελφοι, για την Και τώρα, κλείνοντας την διαδικασία Catch the Eye, η συνάδελφος του Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όταν σκέφτομαι την Ουγκάντα, όταν σκέφτομαι πόσο έχει υποφέρει αυτή η υπέροχη χώρα από την εποχή του Αμίν, όταν σκέφτομαι την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θέλω να ευχαριστήσω συναδέλφους που εξέτασαν το θέμα και μας προσήλξαν την προσοχή. Η, το μίσος, η γλώσσα του μίσους, κοιτάξτε που οδηγεί, ξεκίνησε από μια φυλάδα που δημοσίευσε τα στοιχεία που αφορούσαν τον κύριο Κέιτο και τελικά οδήγησε αυτό στο φόνο. Υπάρχει όμως και η γλώσσα του μίσους και εδώ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει στο σελίδα Red Watch. Δημοσιεύει στοιχεία και διευθύνσεις ανθρώπων με εναλλακτικό σεξουαλικό προσανατολισμό, θρησκεία ε, ή φιλετική καταγωγή και καλή την έκφραση μίσου κατά αυτών των μειονοτήτων αυτή στο σελίδα. Πρέπει να σεβόμαστε ανθρώπινα δικαιώματα, όχι μόνο αλλού, αλλά και εδώ στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε την συνάδελφο του Μούνσταν και τώρα ολοκληρώνεται η διαδικασία κραυστία και τώρα να δώσουμε το λόγο στον Επιτρόπο Κάλλας. President, honorable members. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Να ξεκινώ να απολύσω φόρο τιμής στη μνήμη του David Κάτο. Ήταν ένας θαραλέος υποστηρικτής ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ως ηγέτης ε, των ε, LGTB η ζωή του ε, βρισκόταν απειλή το μάλλον και Δυστυχώς στις 15 Νοεμβρίου η εφημερίδα Rolling Stone αυτή η φυλάδα δημοσίευσε τις, ε, τις φωτογραφίες ε, και τα διευθύνσεις αυτών των ε, ατόμων ήταν επιτυχία το ότι κέρδισε την προσφυγή κατά της εφημερίδας. Αυτή ήταν η τελευταία επιτυχία. Στις 22 Ιανουαρίου ο Ντέιβιτ Κάτο δολοφονήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των εκπροσώπων της στην Ουγγάντα ζήτησε από τις αρχές της να ερευνήσουν τον θάνατο του Κέιτο αλλά και να διωχθούν για να, να προσαχθούν στη δικαιοσύνη οι ένοχοι. Θα πρέπει επίσης να μας θυμίσει ο θάνατός του ότι μάλλον το πόσο πάσχουν ε, τα άτομα αυτά, διεμφυλικοί, και λοιπά στην Ουγγάντα και όχι μόνο. Ε, ε με ιστοσελίδα Red Paper ε, αναφέρθηκε στο ζήτημα αυτό. Η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα δικαιώματα των LGTB είναι σαφής. Η ποινικοποίηση της, της πρέπει να καταδικαστεί. Χρειάζεται επίσης ε, να λάβουμε υπόψη την ε, απόφαση 18 Νοεμβρίου 2008. Εμείς ζητήσαμε επανειλημμένα από την κυβέρνηση της Ουγγάντας σε ανώτερο επίπεδο στον πρόεδρό της, δηλαδή και στον Πρωθυπουργό αλλά και στον Υπουργό Δικαιοσύνης να φροντίσουν να σεβαστούν τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων. Ζητήσαμε επίσης να υπάρξει μια αναθεώρηση της νομοθεσίας σε ό,τι αφορά τις μειονότητες και ειδικά τους LGTB. Στις 2 Φεβρουαρίου η Αντιπροσωπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εκπροσώπους των κρατών μελών ζήτησε να εφαρμοστούν οι αρχές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να προστατευτούν ε, οι υποστηριχτέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να εκφράζει τις ανησυχίες της σχετικά με την ομοφοβική συμπεριφορά και ε, ζητούν να προωθηθεί ο διάλογος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης θα συνεχίσει να υποστηρίζει τα οργανώσει ε, προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, η Προσωπία της Ευρωπαϊκή Ένωσης θα συναντηθεί με οπαδούς ε, και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Επιτρόπο Κάλλας και κλείνοντας να αναφέρουμε ότι έχουμε έξι ε, ψηφίσματα και θα κάνουμε κατευθείαν την ψηφοφορία. Περνάμε στο πρώτο θέμα.